αλλά προ όφελο και των τριών θεσμικών οργάνων τη Ένωση, σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Και ευχαριστώ την Κομισιόν για το πνεύμα συνεργασία που έδειξε. Ευχαριστώ όλοι οι πρόεδρο. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Ψηφοφορία θα γίνει στις... την Τετάρτη στι 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, αξιότιμοι συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο θέμα τη ημερησία διάταξη. Προφορικέ ερωτήσει για προφορική απάντηση από την Κομισιόν όσον αφορά τη μεταφορά δεδομένων από τα κράτη-μέλη προ τη ΣΥΠΑ βάσει του μνημονίου συνεννόηση. Υπάρχουν επενδύσεις από την άλλη, την ΚΟΕ και την ομάδα των Προσύνων. Οι υποβάλλοντε, Η κυρία Ινφέλ πρώτα. Yes, thank you. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μπορώ να είμαι πολύ σύντομη. Νομίζω ότι η προφορική ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Επί του παρόντος, επεξεργαζόμαστε μία δέσμη για τα στοιχεία που αφορούν τους επιβάτες PNR. Έχει προετοιμάσει και ένα σχέδιο για τις διαπραγματεύσεις με τον Καναδά, την Αυστραλία και τη ΣΥΠΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, στο μεταξύ, τα κράτη-μέλη διαπραγματεύονται διμερώς με τις ΙΠΑ την ε, μεταφορά προσωπικών δεδομένων ή μάλλον ε, σε ό,τι αφορά την παροχή πρόσβασης ε, στις ΙΠΑ σε ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων που έχουν να κάνουν και με στοιχεία επιβατών πριν τοποθετηθεί το Κοινοβούλιο για οποιαδήποτε πρόταση σχετικά με το PNR ή η συμφωνία PNR, θα πρέπει να γνωρίζουμε πώ έχει κατάσταση. Διότι αν τα κρατημέλη συμφωνούν διμερώς με τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, να μεταφέρουν στοιχεία PNR, διερωτώ με εγώ τι κάνουμε εμείς εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο. Επίσης ε, μου είπαν, αλλά δεν μπορούμε να το επαληθεύσουμε σε καμία περίπτωση, γιατί είναι μυστικές αυτές οι διμερείς συμφωνίες και διαπραγματεύσεις, ε, Ίσως πάντως πρόκειται να αφορούν στοιχεία PNR για ε, υπηκόους τρίτων χωρών, όχι ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ε, πολιτών που πηγαίνουν σε άλλους προορισμούς και όχι προς τη ΣΥΠΑ και ίσως να μην καλύπτονται από πιθανές συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ύπα. Πρέπει λοιπόν αυτό να διευκρινιστεί πρωτού συνεχίσουμε τις συνομιλίες για το PNR. Και τέλος, κύριε Επιτροπέ, το Σαββατοκύριακο κατά τύχη ενημερώθηκα για κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που λέγεται One Stop Security. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται ε, με την ε, αρμόδια για την ασφάλεια των μεταφορών αρχή στις Ηνωμένε Πολιτείε. Και αφορά τις μεταφορές, ε, τις μετακινήσεις πολιτών από και προς ΗΠΑ και τους ελέγχους ασφαλείας όταν ταξιδεύουν Ευρωπαίοι πολίτες στην Ευρωπαϊκή, ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη ΣΥΠΑ, οι έλεγχοι ασφαλείας γίνονται όλο και πιο αυστηροί αλλά διαπραγματεύεται ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ελάφρυνση των ελέγχων ασφαλείας για τους Αμερικανούς που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ξέρω και θα ολοκληρώσω με αυτό ότι εάν συμβαίνει αυτό, αν οι ΙΠΑ είναι αυτές οι οποίες έχουν επιβάλει αυτά τα πρότυπα ασφαλείας, ε, θέλω να ξέρω πώς, ε, πώς θα συνεχίσουμε αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Σίπελ για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα αναφερθήκαμε συχνά σε συνδίκη της αγώνης και θέλω να πω κάτι θετικό σχετικά. Οι περισσότεροι πολίτε τη Ευρώπη θεωρούν ότι είναι καλό που μπορούν να ταξιδεύουν χωρί να σταματάνε στα σύνορα στην Ευρώπη, ότι μπορούμε να κινηθούμε ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμω σημαίνει ότι αφήνουμε και κάποια ίχνη στοιχείων προσωπικών. Γιατί τα προσωπικά στοιχεία δεν είναι πια σε ένα κράτος μέρος μόνο, αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό είναι καλό και στον με αυτό που πρόκειται για την προστασία των προσωπικών στοιχείων Ευρωπαίων πολιτών να έχουμε περισσότερες αρμοδιότητες στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί οι πολίτες δικαίω αναμένουν τα στοιχεία τους να προστατεύονται σωστά σε όλη την Ευρώπη και να μην μεταφέρονται περιτά πολλά στοιχεία ενδεχομένω και σε τρίτες χώρες. Πώς μπορούμε εμείς όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το λέω ξεκάθαρα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μαζί με τα κράτη-μέλη δηλαδή να εξασφαλίσουμε αυτή την προστασία όταν αφενός η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει τις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες για την μετάδοση των στοιχείων ε, το πού θα χρησιμοποιηθούν ποιοι είναι οι μηχανισμοί προστασίας που χρειάζονται για τα στοιχεία αυτά και ταυτόχρονα με μονομένα κράτη-μέλη διαπραγματεύονται με τρίτες χώρες για στοιχεία που δεν αγνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε ποια στοιχεία είναι, ποια είναι τα πρότυπα προστασίας, κατά πόσον τα στοιχεία διπλά μεταφέρονται ή μεταφέρονται κάποια στοιχεία προσωπικά που εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακριβώς δεν επιτρέπουμε να μεταδοθούν. Και κάτι άλλο που ίσως δεν το έχουν κατά νου τα κράτη-μέλη. Εάν ένα κράτος μέλος διαπραγματεύεται με μια τρίτη χώρα, πώς μπορώ να εξασφαλίσω, πώς μπορεί το κάθε κράτος μέλος να το εξασφαλίσει, μπορεί να το εξασφαλίσει. Ότι εάν προωθούνται, προωθούνται μόνο στοιχεία δικών του πολιτών. Γιατί έχουμε αυτή την, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δει να συλλέγονται κεντρικά στοιχεία πολιτών από διάφορες χώρες μέλη και στα οποία έχουν πρόσβαση διάφορες χώρες. Δηλαδή, πάει κάποιο, πάω εγώ σε μια χώρα που συλλέγει τα δική μου στοιχεία και η, χώρα αυτή αποφασίζει να προωθήσει τα δικά μου στοιχεία σε κάποιον άλλο. Δεν επιτρέπεται αυτό όμως. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα νέα ειδικά βάρη των θεσμικών οργάνων και να τηρούν τους κανόνες. Δηλαδή η προστασία των δεδομένων είναι και θέμα ευρωπαϊκό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να φροντίσουμε ο μικρότερο δυνατό αριθμό στοιχείων να προωθείται και για πάρα πολύ συγκεκριμένου στόχους. Και αυτό να μην καταστρατηγείται από διμερεί συμφωνίε. Ευχαριστώ. Κύριο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το τελευταίο χρόνο, συνάδελφοι, επανειλημμένα συζητήσαμε διάφορα θέματα που αφορούσαν την προστασία των δεδομένων, την ιδιωτική ζωή επίσης των Ευρωπαίων πολιτών, για να εγγυηθούμε τη φυσική ασφάλεια των πολιτών που ταξιδεύουν αεροπορικώς, μας λέγουν ότι θα πρέπει να δίνουμε κάποια από τα προσωπικά τους στοιχεία. Αυτό βέβαια έχει και πολιτικές και νομικές επιπλοκές και συνέπειες. Αν συμφωνήσουμε για αυτή την ανταλλαγή στοιχείων, ξέρουμε ότι όποτε προκύπτει κάποιο πρόβλημα, προσπαθούμε να το επιλύσουμε. Ξεκινήσαμε με το SWIFT και τώρα έχουμε το PNR. Αλλά δεν ξεκινάμε από την αρχή, από το μηδέν θα πρέπει να δούμε πώς προστατεύουμε τα στοιχεία και να εφαρμόσουμε σχετικές διατάξεις παντού με όλους τους διεθνείς εταίρους μας. Είτε είναι η η Σαουδική Αραβία, η Κίνα, η Νότια, η Νότια Κορέα στο μέλλον. Θα υπάρχουν και άλλοι διεθνείς εταίροι που θα ζητήσουν στο μέλλον τέτοια στοιχεία. Λοιπόν, Εάν κινούμεθα κατακαιρματισμένα θα δημιουργηθεί δύσκολη κατάσταση. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει την περίπλοκη εικόνα να τη δει στο σύνολό της είναι η ίδια η κατάσταση κακή και θα χειροτερεύσει αν τελικά διαπιστωθεί ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν υπογράψει υπομνήματα συμφωνίας με τις ΗΠΑ σχετικά ε, με την μετακίνηση ε, επιβατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που μεταβαίνουν στις ΗΠΑ. Είναι σημαντικός εταίρος η ΗΠΑ, δεν λέω αξιοθαύμαστη χώρα από πολλές πτυχές και έχουμε κοινέ αξίες, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αν τα κράτη-μέλη επιτρέπουν την υπονόμευση των διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσης στο σύνολό της είναι μια θέμητη προσέγγιση αυτή από πλευράς αυτών των κρατών μελών και μπορεί να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις και με τη ΣΥΠΑ, αλλά να υπονομεύσει και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θα γίνει πιο δύσκολο στο μέλλον να πετυχαίνουμε την προστασία των δεδομένων που θέλουμε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε αν διαπραγματεύεται σήμερα ξεχωριστά με τα κράτη-μέλη, ε, πού θα σταματήσει, μπορεί στο μέλλον να διαπραγματεύονται οι ΗΠΑ με, με διάφορε αεροπορικέ εταιρείε για την ε, διαβίβαση των στοιχείων επιβατών όταν κλείνουν εισιτήριο. Κάποιο πρέπει να προασπιστεί τελικά τα δικαιώματα των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Το Κοινοβούλιο προσπαθεί να το κάνει αυτό. Είναι σημαντικό και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τα κράτη-μέλη, οι ΗΠΑ να καταλάβουν και να αναγνωρίσουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να πατήσει φρένο, να πατήσει το κόκκινο κουμπί όσον αφορά το PNR Έχουμε δικαιώματα, πρέπει να υπερασπιστούμε, μπορούμε να απορρίψουμε διεθνείς συμφωνίες, όπως κάναμε και με το SWIFT, αν δεν πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις και δεν παρέχεται το επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων των πολιτών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άλμπρεχτ για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας κυρίες και κύριοι της Επιτροπής, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να σας βάλετε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη αυτή την ερώτησή μας. Τώρα έχει ένα θέμα αρχής, δηλαδή κατά πόσον ε, έχει νόημα να εργαζόμαστε πάνω σε διατάξεις για την προστασία των δεδομένων όταν ταυτόχρονα πίσω από την πλάτη μα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο αλλά και ίσω πίσω από την πλάτη των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, διαπραγματεύονται ε, συμφωνίε που υποσκάπτουν αυτά τα πρότυπα. Η διατλαντική συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική, ιδίω για τη δημιουργία ενό χώρου ελευθερία και δικαίου. Αυτό δεν επιτρέπεται όμω στο τέλο να οδηγήσει στην ε, προάσπιση συλλογικών δικαιωμάτων καταπατώντας τα ατομικά δικαιώματα. Και αυτό είναι ένα θέμα της ε, προστασίας των ε, προσωπικών δεδομένων στη διεθνή συνεργασία και είχαμε πολλές φορές στο παρελθόν ότι οπωσδήποτε είτε όταν πρόκειται για θέματα των στοιχείων των αξιωτών είτε για την πρόσβαση σε τραπεζικά στοιχεία θα πρέπει να υπάρχει ένα δίκαιο που να μπορεί να εφαρμοστεί ατομικά και μεμονωμένα. Δεν γίνεται όμως αυτό και γι' αυτό είπαμε ίσως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα ότι θέλουμε γενικά πρότυπα που να εφαρμόζονται παντού και να ισχύουν και για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Εγώ όσον αφορά τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ έχω να πω ότι αυτό ε, ισχύει όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διμερεί συμφωνίε με τη ΣΥΠΑ. Καλό είναι αυτό, αλλά δεν πρέπει να οδηγήσει στο να υποσκάπτονται τα πρότυπα που έχουν συμφωνηθεί από την Ένωση με τη ΣΥΠΑ, περί αυτού πρόκειται, και ταυτόχρονα θα πρέπει να παραμείνουμε μέσα στα πλαίσια του ισχύοντος δικαίου με τη συνθήκη της Λισαβόνας ασχολείται με το θέμα αυτό δικαίως όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά έχουμε ταυτόχρονα ένα πλαίσιο δικαίου που λέγεται ότι όταν υπάρχει μια συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παραδείγματο κάνει τα στοιχεία των δεξιωτών, τότε δεν μπορούν πια οι χώρε μέλη να διαπραγματευτούν πέρα αυτού. Και γι' αυτό σας καλώ να παρέμβετε προς τα κράτη-μέλη και εσείς ε, από την Κομισιόν και η Προεδρία του Συμβουλίου να σταματήσουν αυτές τις διαπραγματεύσεις και επίσης να τηρήσουν την βάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι σαφές για μας το Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μία φωνή στις διαπραγματεύσεις αυτές. Και αυτή η βασική αρχή θα πρέπει να τηρείται. Μία φωνή με την οποία θα διαπραγματεύουμε και όχι συνεχή διαπραγματεύσει σε διμερές επίπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Άλμπρεκτ. Εξ ονόματο της Επιτροπής η κυρία Δαμανάκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. I very much welcome the questions of χαιρετίζω τα ερωτήματα των βουλευτών και θα πρέπει να πω ευθύ εξ αρχή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται την ευαισθησία σα για την προστασία των δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα λοιπόν ε, και να το πιάσω από την αρχή. Θα γνωρίζετε φαντάζομαι ότι τον Αύγουστο του 2007 εξυγχρονίστηκε το πρόγραμμα κατάργησης ε, της απέτηση για θεώρηση διαβατήριου από τις ΗΠΑ. Στόχο ήταν ναι, βέβαια και η βελτίωση τη ασφαλείας. Σίγουρα επηρεάζονται εξίσου όλα τα κράτη-μέλη. Είτε είναι στο πρόγραμμα Visa Waiver είτε όχι. Και ε, μια χώρα μπορεί να παραμείνει ή να μπει σε αυτό το πρόγραμμα εάν συμφωνήσει να συνεργάζεται με τις Ηνωμένε ε, Πολιτείες για θέματα επιβολής ε, του νόμου. Έτσι έχουν τα πράγματα. Συγκεκριμένα χρειάζεται ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με θέματα επιβολής ε, του νόμου. Αυτός ο νέος νόμος οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει μια διτή διαδικασία όπως είπατε. Από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε διαδικασία μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με προποθέσει ε, πρόσβαση ε, στο πρόγραμμα Visa Waiver των ΙΠΑ σε ό,τι αφορά θέματα που εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή Αρμοδιότητα και είχε να κάνει με την πολιτική επιστροφή επικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ασφάλεια ταξιδιωτικών εγγράφων, ασφάλεια αερολιμένων. Αυτά τα ζητήματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μα, στην ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Τώρα, υπάρχει δεύτερη διαδικασία, η διμερή διαδικασία, που εξακολουθεί να ισχύει μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών και ΕΠΑ. Και αυτό για να ικανοποιηθεί το αίτημα της Ευρωπαϊκής, των ΗΠΑ για συνεργασία σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την ε, ασφάλεια. Όσα κράτη-μέλη δεν είναι μέλος του προγράμματος VisaWare θα πρέπει να ε, πληρούν αυτού του προποθέσει πρώτα απ' όλα και μετά να ενταχθούν στο πρόγραμμα για την κατάργηση τη βία. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μα. Όσα κράτη-μέλη είναι ήδη σε αυτό το πρόγραμμα, οι διαπραγματεύσει αυτέ θα γίνουν σε μεταγενέστερο στάδιο. Επομένω, για τα κράτη αυτά τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Με βάση τι πληροφορίε που συγκέντρωσε από τα κράτη-μέλη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι ο μόνο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Οκτώ κράτη-μέλη έχουν υπογράψει μνημόνια συνεννόηση με τι Ηνωμένε Πολιτείες, τα οποία αναφέρεται ότι συμφωνούν να συνεργάζονται με τις Ηνωμένε Πολιτείες για αυτά τα ζητήματα. Πρόκειται για την, την Τσεχία, την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Λετωνία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα και τη Σλοβακία. Με τον τρόπο αυτό και αυτό ήταν το πρόβλημα που προσπαθεί να επιλύσει αυτή η διαδικασία. Αυτά τα, κράτη, τα οκτώ κράτη μπόρεσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Visa Waiver. Γι' αυτό έγιναν αυτές οι συμφωνίες τελικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλαβαίνει ότι τα μνημόνια συνεννόησης δεν είχαν ε, στόχο να αποτελέσουν ε, βάση νομική βάση ανταλλαγής ε, δεδομένων μεταξύ ΙΠΑ και αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Πρόκειται απλά για έκφραση της πρόθεσης των δύο πλευρών να έχουν ειδικέ ρυθμίσεις, συμφωνίες που θα διέπουν την ανταλλαγή δεδομένων. Περί αυτού πρόκειται. Πρέπει να υπογραμμίσω το εξή. Οι πληροφορίες για το ακριβές περιεχόμενο των μνημονίων συνεννόησης είναι στη διάθεση των κρατών μελών. Αυτά, αυτοί έχουν τα στοιχεία. Όπω, παραδείγματο χάρη, κατηγορίε δεδομένων που διέπονται από τα μνημόνια. Επομένω, εάν θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει να τις αναζητήσει στα οικία κράτη-μέλη. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και έρχομαι τώρα στις δικές μας ευθύνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εξασφαλίσει ή είπα να μην ζητούν διμερεί ρυθμίσει και διευθετήσεις με τα κράτη-μέλη για την ανταλλαγή στοιχείων PNR. Of PNR data, since this was a... Καθότι αυτό το ζήτημα εμπίπτει στην ευρωπαϊκή αρμοδιότητα με βάση τη συμφωνία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη ΣΥΠΑ για τα στοιχεία PNR. Αυτό κάναμε. Τέλο, στι διαπραγματεύσει για τη συμφωνία ΕΠΑ Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε μια ανταλλαγή αλληλογραφία για να καταγραφεί το ότι οι νόμικε απαιτήσει των ΕΠΑ για τη συνεχιζόμενη ε, συμμετοχή στην συμφωνία αυτή πρέπει να πληρούνται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε σαφές ότι η ανταλλαγή αυτή επιστολών που συνεχίζεται μαζί με τις διαπραγματεύσεις δεν θα μπορούσε να δώσει πρόσβαση βάσει δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα οι ομιλητές εξ των πολιτικών ομάδων. Πρώτο ο κύριος Κοέλιο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφε, κυρία Επίτροπε. Άκουσα τις απαντήσεις σας και κάπως όμως ε, μπερδεύτηκα. Γιατί μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη μία πλευρά ότι αν θέλουμε περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να χτυπήσουμε την πόρτα των κρατών μελών. Ο μόνος τρόπος που μπορούμε αυτό να το αντιληφθούμε είναι ως εξή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι δεν έχει μέσο να πείσει τα κράτη και να τα πιέσει σε αυτή τη φάση. Και μετά ακούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τις Ηνωμένε Πολιτείες να μην παρέχουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις συμφωνίες μας με την παροχή δεδομένων. Τι μπορεί να είναι πιο εύκολο από το να έρθει σε επαφή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα κράτη-μέλη να το διελευκάνει το θέμα. Λοιπόν, ένα πράγμα θα πρέπει να διαπιστώσω ότι έχει κάποια δυναμία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τοποθετηθεί ε, σωστά ανησυχεί το Κοινοβούλιο σαν αυτό το θέμα. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, ένα τιμωρησία διαιρούν για να βασιλεύουν. Και λυπούμεθα διότι κάποια κράτη-μέλη αποφάσισαν να επιλέξουν διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ παραβιάζοντας κάθε έννοια αλληλεγγύης ευρωπαϊκής. Όμως υπάρχει μια λογική απέκτηση των ευθυνών από πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που δεν δίνουν δύναμη διαπραγμάτευση στην Ευρώπη. Δεν μιλά Ευρώπη με μια φωνή. Θα πρέπει να φροντίσουμε ούτω ώστε μέσω διμερών συμφωνιών να μην υπάρχει πρόσβαση στι βάσει δεδομένων. Και θα πρέπει τα μυστικά που καλύπτουν αυτέ τι διαπραγματεύσει να μην οδηγούν στο να μην ενημερώνουν τα εθνικά κοινοβούλια, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει τι πληροφορίε όσον αφορά τα θέματα. Σωστά λοιπόν εμείς ανησυχούμε. Είναι ανησυχίες που δεν καθησυχάστηκαν από αυτά που μας είπε η κυρία Επίτροπος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μέλτσερ για ένα λεπτό. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. I'm sorry, I'm sorry, Mr. Μέλτσερ. Ο κύριος Άλβαρο πρώτα για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επίτροπο που απάντησε με τον συναδέλφους ε, κυρίας Μάλστρομ αλλά νομίζω ότι έχουμε διαφορετική βάση εργασίας γιατί δεν πρόκειται μόνο για το θέμα των ε, στοιχείων PNR. Ε, ελέγχθη ξεκάθαρα ότι υπάρχουν διακτηρικά αποτυπώματα ποινικού μητρώου, ε, DNA και όλα αυτά με το σύστημα που εμείς έχουμε πετύχει με την συνθήκη της Ρώμης. Αυτό είναι θέμα της ευρωπαϊκής πολιτικής Πραγματικά αυτό είναι πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε, να βρούμε πώς θα μπορεί να γίνει, να το συζητήσουμε κλπ. Αυτό που με ανασυχίζει είναι ότι ούτε η Κομισιόν ούτε το Συμβούλιο έχουν το θάρρος να πούνε στις είπα ως εδώ και με παρέχει. Παρέχει. Δεν μπορούμε να ε, εκμεταλλευτούμε την ε, απελευθέρωση από τη θεώρηση, το Visa Waiver, προς μια χώρα όπω η Αυστρία πούμε, να της πει ότι εμεί θα σας αφαιρέσουμε το δικαίωμα αυτό αν δεν κάνετε αυτό που θέλουμε. Γιατί η συμφωνία λέει ότι εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση δίνουμε αυτή την ε, απελευθέρωση στη ΣΥΠΑ. Λοιπόν, εμείς θέλουμε τη ε, διατλαντική ε, συνεργασία και εταιρική σχέση. Αλλά θα πρέπει όμως να είναι επικοδομητική η σχέση αυτή. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να κατεύθυνση αυτή και το ίδιο περιμένουμε και από του Αμερικανού πολίτες και από την Αμερικανική πολιτική. Και ελπίζει η Κομισιόν και το Συμβούλιο να το τονίσουν αυτό πολύ περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Äh, Πρόεδρε, και τότε που είχαμε προετοιμάσει την, ε, το συμβασμό SWIFT ήταν σαφές αυτό, αυτό που θεωρείται ότι ήταν προστασία των περιοριστικών δεδομένων ήταν μια γεωγραφία Και τώρα είναι ξεκάθαρα. Το κοινοτικό πρόγραμμα επιτήρησης δεν αποδείχθηκε αναποτελεσματικό σε μερικά χρόνια, αλλά σε μερικού μήνες όλες οι συμφωνίες που υπάρχουν καταδεικνύουν ότι οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται για εταίρους αλλά εκείνους που λένε ναι και αμήν σε όλα που κάνει η Αμερική. Η ΕΠΑ πολλά χρόνια μπορούσε να έχει ε, ε, πρόσβαση στα τραπεζικά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν ε, θεωρήθηκε ότι θα υπάρχει ένας Ευρωπαίος ελεκτής, από την πίσω πόρτα είπα πάλι μπορούν να το κάνουν. Εγώ ε, θα θεωρώ ότι θα πρέπει να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης με τις διαθεμικές συμφωνίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Στράσερ για δύο λεπτά. Αξιότιμη κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, όπως είπε και κάποιος προλαλής σας, θα πρέπει πραγματικά να αναγνωρίσουμε ότι ήρθαμε εσείς σε εδώ και κάνετε μια δήλωση. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι το δικό σας θέμα αυτό, αλλά από την άλλη μεριά λέω ξεκάθαρα ότι η δήλωση της Κομισιόν δεν μας εικονοποιεί καθόλου. Γιατί έγινε κάτι που σας παρακαλώ να σημειώσετε. Όλες οι σημαντικές πολιτικές ομάδες εδώ στο σώμα θέλουν να συζητήσουν επί τις και ενοχλούνται φοβερά όταν βλέπουμε ότι δεν δράει η Κομισιόν. Το ίδιο έγινε και με τη συμφωνία SWIFT. Στην περασμένη σύνοδο επιστήσαμε την προσοχή της Κομισιόν στα 14 δολάρια τέλος εισόδου και τώρα πάλι λέμε τι κάνει η Κομισιόν, τι κάνει το κράτη-μέλη και τώρα ακούω ότι υπάρχει συζήτηση για ε, προτιμησιακές θέσεις των μεγαλών είναι των Ευρωπαίων. Θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι εδώ θέλουμε να συζητήσουμε πολύ σοβαρά με την Κομισιόν για τα θέματα αρχής και θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει αμοιβαιότητα. Δηλαδή, όχι να υπάρχει πρόσβαση σε ε, στοιχεία από την Ευρώπη, αλλά θα πρέπει αυτή η διαδικασία, ας πούμε, που να μην συνεχίσει να πούμε τι γίνεται με τα δικαιώματα των πολιτών. Ο πολίτης έχει δικαίωμα να ξέρει ποια από τα στοιχεία του χρησιμοποιούνται πού και πώς. Και οπωσδήποτε όλα αυτά θα πρέπει να βασίζονται σε ευρωπαϊκή βάση. Αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η Κομισιόν επιδίνωσε τη διαπραγματική τη θέση με τους Αμερικανούς γιατί δεν συντονίζεται με τα κράτη-μέλη και γιατί η ίδια δεν δρά. Πότε θα αρχίσουν αυτές τις διαπραγματεύσεις, πότε θα δούμε να υπάρχει κάποια δραστηριότητα το SWIFT προχώρησε με την πίεση του Κοινοβουλίου σε ένα μήνα. Για ίδιες δραστηριότητες χρειάζομαι για τα PNR και για τα γενικά στοιχεία. Ευχαριστώ. Στη διαδικασία του ΚΑΤΣΤΙΑΙ, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε τρεις ε, ομιλητές. Ε, πρώτα, I'm sorry, Sophie, it's Eye afterwards. What, what? I can't give the floor now. If it's, if it's a point of order, yes. If it isn't, no. Unless you want to be in the catch the eye, I can consider that. Αν θέλετε κάποια διευκρίνηση μετά το catch the eye. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία με αποτελεσματικότητα. Αυτό δεν είναι εφικτό αν δεν υπάρχει διεθνή συνεργασία στον τομέα αυτό. Πρέπει βέβαια να τηρούνται και οι δημοκρατικοί κανόνες εν των του Ατλαντικού. Στι διμερεί τώρα συμφωνίε μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη φαίνεται να προχωρούν. Οι διαπραγματεύσει όμω βασίζονται μόνο στα εθνικά κοινοβούλια. Οι διάφορε συμφωνίε που αναφέρθηκαν ζητούσαν όμω δημοκρατικό έλεγχο και διαφάνεια. θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ε, και τι ανησυχίε τη κοινή γνώμη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαβίβαση ορισμένων δεδομένων, ε, εγώ δεν θα είχα ιδιαίτερο πρόβλημα. Θα πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ αυστηρό έλεγχος όμως ε, και θα πρέπει κάποιοι βουλευτές και δικαστές να έχουν και αυτοί ένα λόγο σε αυτή την ιστορία. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία των πολιτών, πρέπει να πω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα και όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνία των πολιτών. Η διαβίβαση στοιχείων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τη ΣΥΠΑ δικαιολογήθηκε από την προσπάθειά μας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της προστασίας της συλλογική ασφαλείας των πολιτών. Βεβαίως αξέπαινος αυτός ο στόχος. Όμως, καμιά φορά, έχω την εντύπωση την άσχημη ότι προς όφελος εις όνομα της καταπολεμής τρομοκρατίας ε, υπονομεύουμε την ιδιωτική ζωή των πολιτών μας. Ε, που δεν θα ήθελα να υπονομεύσω τι διαπραγματεύσει μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ενώσεω και είμαι πεπισμένη ότι οι ΗΠΑ είναι ο πιο στενό και ισχυρό σύμμαχό μα. Αλλά το ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται δημερό με κράτη-μέλη, αυτό το γεγονό ότι διαπραγματεύονται τα κράτη-μέλη και όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη, αυτό έχει δημιουργήσει καχυποψίε και για να υπερασπιστώ τις χώρες που υπέγραψαν αυτά τα υπομνήματα συνεννόησης. Θα τις υπερασπιστώ. Αυτά τα κράτη-μέλη δεν ήταν μέλη του προγράμματος Visa Waiver. Και θεωρήσαμε ότι έπρεπε να βρούμε αυτή τη λύση. Στο μέλλον θα εκπροσωπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη-μέλη. λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, είμαι πεπισμένο ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τι προσπάθειε για την καταπολέμηση τη τρομοκρατίας που εξακολουθεί να απειλεί τον πολιτισμένο κόσμο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χειρισμό προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων ταξιδιωτών ε, υπό το πρόσχημα τη καταπολέμηση τη τρομοκρατίας, ε, φαίνεται ότι πάσχει από έλλειψη συντονισμού ή είπα από την πλευρά τους συλλέγουν ε, τα στοιχεία για τους Ευρωπαίους πολίτες με βάση συμφωνίες με τα κράτη-μέλη μεμονωμένα, με διμερείς συμφωνίες δηλαδή, και με βάση συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι πλέον, δεν θα πρέπει να είναι πλέον αποδεκτή αυτή η διτή, αυτή η διπλή διαδικασία. Θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση κατά τρόπο ώστε να μην επιτρέπεται να παραβιάζονται τα δικαιώματά μας και να παρακάμπτονται οι νόμιμε διαδικασίε. Θα πρέπει λοιπόν απέναντι στη ΣΥΠΑ να επιμείνουμε για να υπάρχει σεβασμός στις αρχές της αμοιβαιότητα. Και θα πρέπει τα ευρωπαϊκά δεδομένα να μεταφέρονται με βάση κανόνες, τους κανόνες που εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Πήρα, δέχτηκα κυρία Μορβάη σε εξαιρετική περίπτωση. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Συνάδελφοι, οι παρεμβάσει του ενό λεπτού είναι κάτι που δεν λειτουργεί τελευταία στιγμή. Αν θέλετε να συμμετέχετε στη διαδικασία, σα παρακαλώ να σηκώνετε το χέρι σα εκ των προτέρων. Κάνω μια εξαίρεση, διότι δεν υπάρχουν πολλοί στον κατάλογο σε αυτή τη φάση. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω, ε, δεν υπάρχει τόσο ζωή και ενδιαφέρον φαίνεται για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το λέω όπως η παράσπιση μου και δεν παίρνω το χρόνο άλλων. Οποιαδήποτε προστασία δεδομένων και σχετική διαδικασία ή αδίποτε διαδικασία που παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα όσον αφορά την προστασία των δεδομένων θα πρέπει να σχετίζεται με συγκεκριμένο στόχο, ξεκάθαρο στόχο και θα πρέπει να μπορούμε να πετυχαίνουμε αυτό τον τεκμηριωμένο στόχο σύμφωνα με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ποια είναι η δικαιολογία, ποιος είναι ο στόχος ο δικαιολογημένο, ο τεκμηριωμένος και πώς η διαβίβαση προσωπικών στοιχείων μπορεί να πετύχει τον εν λόγω στόχο. Με άλλα λόγια, πώς θα χρησιμοποιήσουν οι Αμερικανοί αυτά τα στοιχεία. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που απευθύνω προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το άλλο ερώτημα, γιατί χρησιμοποιούν δύο διαφορετικά επίπεδα ελέγχου έναντι των παλαιών και έναντι των νέων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένη τη χώρα μα τη Ουγγαρία. Γιατί ένα Ούγγρο πολίτη είναι πιο επικίνδυνο από την έποψη τη τρομοκρατία από οποιονδήποτε πολίτη παλαιότερων κρατών μελών. Αυτό ήταν ένα θέμα που ετέθη κατά τι διαπραγματεύσει ή πρόκειται στο μέλλον να είναι θέμα. Ευχαριστώ. Θέλω μια διευκρίνηση επί δύο σημείων εξεπλάγει κάπω, ακούγοντα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λέγει ότι το θέμα του προγράμματο Visa Waiver επηρεάζει μόνο τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι αυτό είπατε. Ενώ το 2007 ρω αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πει ότι είχε την αποκλειστική αρμοδιότητα στον τομέα και θα έπρεπε να παραχωρήσει αρμοδιότητα στα κρατη μέλη ενδεχομένω. Τώρα πώ να το εκλάβω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άλλαξε άποψη όσον αφορά τι αρμοδιότητε που διαθέτει. Δεύτερον, προ διευκρίνηση, κυρία Επίτροπε. Είπατε ότι δεν γίνεται καμία αμνία στα, στη μεταφορά των στοιχείων PNR στα διάφορα μνημόνια. Μπορώ να σας δώσω ένα μνημόνιο που αναφέρεται στο PNR. Αυτό σημαίνει ότι η ίδια η Κομισιόν δεν ξέρει τι συμβαίνει. Εγώ θα σας δώσω ορισμένες διασαφηνίσεις Το Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναβάλει τη συζήτηση για δύο συμφωνίες PNR, διότι θεωρούσαμε ότι η Κομισιόν μπορεί να είναι τόσο υπεύθυνη όσο και εμείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αναρωτιέμαι κατά πόσο πρέπει να της δείξουμε εμπιστοσύνη. Ελπίζω να μην μας απογοητεύσετε. Ε, εκ μέρους της Επιτροπής, η κυρία Δαμανάκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορώ Καταρχήν μάλλον θα ήθελα να πω ότι η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά θα ήθελα να κατανοήσετε ότι βρίσκομαι εδώ για να σας δώσω επεξηγήσεις. Δεν μπορώ όμως να ε, δεχτώ αυτά που λέτε ότι η Επιτροπή δεν είναι ευαισθητοποιημένη στην προστασία δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών. Επίσης, δεν αντικαθιστώ μόνο το συνάδελφο χωρίς να γνωρίζω το θέμα και το τι συμβαίνει στην Επιτροπή όλοι μας ξέρουμε τι συμβαίνει επί όλων των θητημάτων και είμαστε ιδιαίτερα ε, ευαισθητοποιημένοι ως προς την προστασία δεδομένων. Τώρα, πρέπει να τηρήσουμε τη συνθήκη της ε, ε, Λισαβόνας ή όχι. Τι θέλετε να αγνοήσουμε το Συμβούλιο. Είναι πολύ εύκολο να λέτε αυτά που λέτε, ότι δηλαδή η ευρωπαϊκή φωνή θα πρέπει να είναι μία και ενία. Συμφωνώ μαζί σας. Τι προτιμάτε όμως να πούμε ότι αγνοούμε το Συμβούλιο ολοσχερός. Θα ήθελα να σας πω, μιλώντας για δεδομένα και όχι όνειρα, ότι ήδη ζητήσαμε από το Συμβούλιο, και αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο, ήδη έχουμε ζητήσει και έχουμε προτείνει από τον προηγούμενο Μάιο στο Συμβούλιο το μελλοντικό, η μελλοντική συμφωνία πλαίσιο Ευρωπαϊκή Ένωση είπα εάν αναφέρεται σε προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να ισχύει και για τα δεδομένα κρατών μελών. Αυτό προτείναμε, επακριβώς αυτό προτείναμε, αυτό που αναφέρατε εδώ και αν συμφωνηθεί τότε θα κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ε, περί αυτού πρόκειται. Αν δεν συμφωνηθεί με το Συμβούλιο, τι, τι, τι, τι, τι μου προτείνετε να κάνω, να πάω στα κράτη-μέλη και να τους πω ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Εντάξει. Αυτή είναι η δική σας πρόταση, κατανοητή η απάντησή μου είναι απλή. Θα πρέπει να τηρήσουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό μπορώ να σας πω. About some other issues, very, very interesting. Ως προς άλλα ενδιαφέροντα ζητήματα, άκουσα για την Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων και τη Βάση Δεδομένων ΠΡΟΥΜ. Θα πρέπει να σας πω ότι τα κράτη-μέλη Ενδεχομένως, αν έχουν μνημόνια συνεννόησης και διμερείς συμφωνίες, μπορούν να δώσουν δεδομένα από τις εθνικές ε, βάσεις δεδομένων, όχι από τη βάση πριν ή την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Και ήμουν σαφής ως προς αυτό. Επίσης είπα ότι ζητήσαμε από τις ΕΠΑ μέσω επιστολών και το διαπραγματευόμαστε αυτό, ότι ζητήσαμε οι διμερείς συμφωνίες να μην αναφέρονται σε στοιχεία PNR. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη δεν διαπραγματεύτηκαν με τις ΙΠΑ διμερώς, αλλά αυτή είναι η θέση της Κομισιόν. Άρα θα ήθελα να πω είναι ότι κατανοώ τις ανησυχίες σας, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε, να διαπραγματευτούμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να προσπαθήσουμε Θεήσουμε να έχουμε δεσμευτικούς κανόνε για τα κράτη-μέλη στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Γιατί αυτό είναι ο μοναδικός τρόπος να επιτύχουμε αυτό που επιθυμούμε. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαπραγματευτεί με τις ΕΠΑ. θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε μια δεσμευτική συμφωνία για τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό μεταβήκαμε στο Συμβούλιο και το παρακαλέσαμε το εξής. Εάν συμφωνηθεί κάτι τέτοιο και εάν μπορούμε να ε, προβούμε σε αυτή τη δέσμευση, τότε θα πρέπει να υπάρχει, να είναι αμφίδρομη η πορεία. Έχετε μια διαφορετική πρόταση με βάση το νομικό πλαίσιο που πρέπει να τηρήσουμε. Εγώ μπορώ να το ακούσω, αλλά αν δεν υπάρχει τέτοια πρόταση θα πρέπει να κατανοήσετε ότι είμαστε πολύ ευαίσθητοι ως προς τα προσωπικά δεδομένα πολιτών και προσπαθούμε να τα προστατεύσουμε. Όμως πρέπει να τηρήσουμε και τη θέση του Συμβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι αυτό το θέμα συνεχίζεται, λαμβάνω υπόψη τις ανησυχίες σας, προσπαθώ να λάβω υπόψη όλα τα στήματα. μπορούμε ως Επιτροπή να μεταβούμε στο Συμβούλιο και να πούμε τι, ότι πρέπει να σταματήσουμε τις συνομιλίες με άλλες χώρες. Μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε. Μπορούμε μόνο να διαπραγματευτούμε και μετά να ε, τους ε, υποδείξουμε να ακολουθήσουμε τη δική μας οδό. Αυτά μπορούμε να πούμε. Κύριε Επίτροπε, επειδή γνωρίζω το θέμα, θα ήθελα να τονίσω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες έχουν εκφράσει μεγάλες ανησυχίες και τώρα ε, βρισκόμαστε στη φάση επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας. Θα πρέπει η Επιτροπή να λάβει υπόψη πολύ σοβαρά αυτές τις ανησυχίες και να μην υπάρχει η αποσύνδεση που υπήρξε στη συμφωνία SWIFT. Επίσης, μιλήσαμε για τις γκρίζες ζώνες που είναι πολύ επικίνδυνες. Εάν κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να δώσει σε τρίτη χώρα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Δεδομένων, ας πούμε στα πλαίσια του Σέγγεν, τότε στο τέλος το τρίτο κράτος μέλος θα μπορέσει να συλλέξει όλα τα στοιχεία στη, της βάσης δεδομένων Σέγγεν που δεν τα παίρνει από τη βάση Σέγγεν αλλά από τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Και υπ' αυτή την έννοια με βάση αυτά που πολύ σωστά αναφέρεται, όπως πολύ σωστά αναφέρεται, θα πρέπει η Επιτροπή με σθένος να προασπιστεί αυτό τον πυλώνα, τον κοινοτικό πυλώνα. Επίσης, θα ήθελα να προχωρήσει αυτό το θέμα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλετε να απαντήσετε, έχετε το λόγο. Συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες τις ανησυχίες και υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αυτό το κατέστησα σαφές εξ αρχής και θα ήθελα να το κατανοήσετε. Αλλά θα θέλαμε στην Επιτροπή να βρούμε ένα νομικό μέσον και τρόπο για να τηρήσουμε τη συνθήκη και να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα δηλαδή να προστατεύσουμε τα δεδομένα προωθώντας το κοινοτικό πυλώνα του θέματος. Αλλά δεν είναι ο μοναδικός πυλώνας που έχουμε. Αυτό θα ήθελα να τονίσω. Θα ήθελα να κρατήσετε, να έχετε κατά νου αυτά που σας είπα και ζητήσαμε και από το Συμβούλιο να δεσμευτεί. Εάν εμείς είμαστε επιτυχής ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων στη δική μας συμφωνία, ζητήσαμε από το Συμβούλιο να δεσμευτεί επί του θέματος. Αυτό είναι ο μόνο, το μόνο νομικό πλαίσιο για να προχωρήσουμε. Έληξε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο σημερινής διάταξη είναι η κοινή συζήτηση σχετικά με την αλληλεία. Η σύσταση του κυρίου Βαλέσα τη Σύμβαση περί της μελλοντικής πολυμερού συνεργασίας στον τομέα της αλληλείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού και η έκθεση της κυρίας Φράγκα Εστέβες «Σύστημα ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της Σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλληλείας